ευχαρίστηση διότι οι προσυπογράφοντες είναι αρκετοί σε σχέση με τις επιστημονικές δυνατότητες της Αφρικής και σε σχέση με τις, την εταιρική σχέση Ευρώπης-Αφρικής και θα ήθελα να ευχαριστήσω και μία ομάδα νέων η οποία ανέλαβε αυτή την συλλογή υπογραφών και να ευχαριστήσω και την κυρία Παντόρ, την Υπουργό της Νοτιού Αφρικής, η οποία θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα για να μας μιλήσει για τη σημασία αυτού του θέματος της επιστημονικής συνεργασίας με την Νότια Αφρική. Θα ήθελα επίσης να παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει θετικά λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αυτής της γραπτής δήλωσης που είναι ύψης της σημασίας όπως σας προείπα για την Αφρική, για την επιστήμη και για τη συνεργασία των δύο υπήρων. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, λοιπόν, στους ε, συντάκτες αυτής της ε, γραπτής δήλωσης. Και τώρα προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη που προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του κ. Ντέιβι σχετικά